και κοινωνικέ συνέπειε μια αποτυχία στην παρούσα φάση θα ήταν πραγματικά ανυπολογίστε. Άρα, επαναλαμβάνω την θέση μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρο, ολοκληρώνεται λοιπόν η κοινή συζήτηση. Αύριο στις 12 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη ε, είναι η δήλωση τη Επιτροπή για το Φόρουμ Ενιαία Αγορά.

Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετωπίζουμε πολλέ φορέ ε, μα οδηγά στο να ξεχάσουμε τον αντίκτυπο στους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν είναι σωστό να κάνουμε μερικά βήματα πίσω για να κοιτάξουμε ποιος είναι ο απότερος στόχος όλων των μεταρρυθμίσεων. Η κοινωνική και η οικονομική ευημερία των ε, συμπολιτών μας. Θα πρέπει να αποδεχτούμε την ευθύνη αυτή για τους ε, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι επίσης καταναλωτές, εργαζόμενοι, εμπειρογνώμονες, αλλά και άτομα που κάνουν αποταμίευση, που ακολουθούν τις επιχειρήσεις τους, είτε είναι μικρές, μεγάλες ή μικρομεσαίες. Και επίσης απασχολούνται στις ε, τοπικές κοινωνίες τους. Όλα αυτά αρκούν για να καταλάβουμε τον αντίκτυπο και τα αλυσιβωτά, τις αλυσιβωτές, αν θέλετε, επιδράσεις. Θα πρέπει να τους δείξουμε ότι η ενιαία αγορά τους δίνει ευκαιρία για ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν ε, διοργανώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στην Κρακοβία με συνεργασία με εσάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Προελληνική Προεδρία ένα φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν 10.000 άτομα και πολλοί φορείς. Θα ήθελα στη παρούσα φάση να ευχαριστήσω την κυρία Ροζοτούν, Μάλκομ Χάρμπορ και τον Σιλμπουμπουσόη, η συμμετοχή των οποίων έκανε το ΣΥΜΦΟ τόσο μεγάλη επιτυχία. Το φόρουμ έκανε, κατέστη δυνατή την ε, συγκέντρωση όλων των φορέων. Μεγάλη επιτυχία, το, η οποία μας οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Μπορέσαμε να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να βελτιωθεί η κατάσταση για πολλούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης και να διακρίνουμε τις ανάγκες τους ε, να ενημερώσουμε για τις μεταρρυθμίσεις που διεξάγουμε. Διαρκώς θα πρέπει να προσπαθούμε να ενημερώνουμε για τις πρωτοβουλίες μας από τη στιγμή που συζητιόνται μέχρι τη φάση της εφαρμογής τους. Τα σχόλια τα οποία συλλέχθηκαν αποτύπωσαν τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της έρευνας για τα 20 ανησυχίες του, του πολίτη ε, της Ευρώπης στην καθημερινότητά του. Η μελέτη επιβεβαίωσε την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης του πολίτη και των επιχειρήσεων και του ρόλου της ενιαίας αγοράς που θα πρέπει να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την αναγνώριση των ε, ε, επαγγελματικών προσόντων, της δημοσίων προμηθειών και γνωρίζουμε ότι η δήλωση της Κρακοβίας που, στην οποία προέβησαν συμμετέχοντας στον φόρουμ είναι σημαντική και είμαστε βιτεθειμένοι να την εφαρμόσουμε. Τρεις ε, βασικές δράσεις διακρίνουμε. Καταρχάς, η ενιαία αγορά να καταστεί ένα πιο ασφαλή τόπο για την καθημερινή δράση του Ευρωπαϊκού του Ευρωπαίου πολίτη. Θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη προς την ενιαία αγορά και να ξέρουν τα δικαιώματά τους όταν κάνουν συναλλαγές σε άλλες χώρες ή όταν μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωπικούς ή επαγγελματικού λόγους. Γι' αυτό θέλουμε να βελτιώσουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αμοιβαίας αναγνωρίσεις για να διευκολύνουμε τον Ευρωπαίο πολίτη και να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν ε, γραφειοκρατικά εμπόδια. Προτείνουμε νομοθεσία για την ε, απόσπαση των εργαζομένων και σε ό,τι αφορά βασικές ελευθερίες που θα δώσουν στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν καλύτερα την ενιαία αγορά. Χτες εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πακέτο μέτρων που σκοπού έχει να διευκολύνει τους πολίτες που μετακινούνται σε, άλλους, σε άλλες χώρες σε ό,τι αφορά επίλυση διαφορών με τους εμπόρους χωρίς απαραίτητα να πάνε στα δικαστήρια θα πρέπει αυτή η νέα μορφή κατανάλωσης να διελευκανθεί. Γιατί σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιείται πολύ περιορισμένα ακόμα. Κατά δεύτερον, η οικονομία της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να καταστεί πιο δυναμική, εφαρμόζοντας πλήρως την οδηγία για τις υπηρεσίες και βελτιώνοντας τα διόδους ε, επικοινωνίας σε άμεση επαφή με τους επιχειρηματίες και συμπεριλαμβάνοντας τους όρους που χρειάζονται για να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί σε μια τέτοια αγορά. Υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένα μέτρα. Η δημιουργία μιας, ε, ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα προωθήσει την ε, κοινοτομία στην ε, Ευρώπη και θα προωθήσει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απλοποίηση των λογιστικών κανόνων, των κανόνων δημοσίων προμηθείων. Και τρίτον, ε, θα αναθερήσουμε τις οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να καταστήσουμε την ε, ζωή και τη δουλειά των εμπλεκομένων φορέων πιο εύκολη και να ε, προωθήσουμε θέματα καινοτομίας. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να πληρώσουμε το νομικό κενό που υπάρχει σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών στην Ευρώπη για να βελτιώσουμε την σχέση μεταξύ των ιδιωτικών αρχών, των δημοσίων αρχών και των ιδιωτικών ε, παροχών. Τέλος, θέλουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε τις σχέσεις μας με τρίτα μέρη για να υπάρξει πιο πολύ αμοιβαιότητα σε θέματα τέτοια δημοσίων προμηθειών. Όλα αυτά τα μέτρα εντάχθηκαν στην, ε, στην πράξη για την ενιαία αγορά και θα πρέπει να εφαρμοστούν. Το 2012 θα είναι καθοριστικό έτος για τη μεταρρύθμιση αυτή. Θα αποτελέσει ένα ορόσημο και το έργο μας για την νέα πρόθεση της ενιαίας αγοράς προκειμένου να σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να εστιαστούμε σε μια νέα ανάπτυξη στο υποτοφό τη δήλωσης τη κρακοβία. Θα διοργανωθούν την εβδομάδα εκείνη ε, εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες και ε, προσδοκώ στη συμμετοχή σας ε, προκειμένου η 20η επέτειο της, της, αγορά να καταστεί επιτυχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα ακούμε τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων με πρώτο ένα διπλό από την Βάδη Βιτεμβέργη, την πατρίδα μου, τον κύριο Σφάπ καταρχάς, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, 3 και 4 Οκτωβρίου το Φόρουμ για την Ιστορική Αγορά στην Κρακοβία γνώρισε πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπως και ο κύριος Δαλή, και σε μια πόλη όχι πολύ μεγάλη, αρκετά μακριά από τις Βρυξέλλες, προσήλθαν όλοι οι φορείς που ενδιαφέρονται για την ιστορική αγορά για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Και προτάσεις για νομοθεσία που ήταν χρήσιμες πιστεύω. Διότι φάνηκε, κύριε Πρόεδρε, ότι σε πολλά θέματα έχουμε σύμπνοια μέσα στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαρτήτως των πολιτικών ομάδων. Με παραδείγματι ενίσχυση των δυνατοτήτων για επίλυση των διαφορών, την ενίσχυση των συνθήκων της προστασίας του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που θέλουμε να προωθήσουμε, την απλούστευση στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι βρίσκουν σύμφωνες όλες τις ομάδες, ε, τις πολιτικές ομάδες και άλλωστε και ο καθηγητής Μόντ στην πρότασή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι χρειάζεται όχι μόνο μια οικονομική διακυβέρνηση αλλά και μια διακυβέρνηση εσωτερικής αγοράς, δηλαδή ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη και για όλους τους εμπλεκόμενους στην εσωτερική αγορά ε, πράγμα το οποίο φυσικά βρίσκει σύμφωνο ολόκληρο το Κοινοβούλιο, πιστεύω. Και έτσι θα ήθελα να φτάσω και στα συμπεράσματα, στα τελικά συμπεράσματα αυτού του Φόρουμ της Εσωτερικής Αγοράς της Κρακοβίας. Ο Υφυπουργό, ο πρώην Υφυπουργό, επεσήμανε πω και τα κράτη-μέλη θα ήταν διατεθειμένα ενδεχομένω να δεχθούν περισσότερε ρυθμίσει εφόσον αυτέ είναι χρήσιμε για την εσωτερική αγορά. Εγώ, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, τη ομάδα μου, θα ήθελα να πω ότι στην ε, ε, διαμόρφωση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ιδιαίτερη αξία αποδίδουμε στο να ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα για ουσιαστική λειτουργία των κανονισμών με διαδικασίες ταχύτερες φυσικά και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει σωστές επιλογές στην υπόθεση αυτή και απλούστευση της, ε, του γραφειοκρατικού φόρτου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σφαπ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Το φόρουμ στην Κρακοβία όντω χαρακτηρίστηκε με μεγάλη επιτυχία. Και πρέπει να επαναλαβούμε αυτό το, αυτή τη διαπίστωση, γιατί πρέπει ό,τι γίνεται καλά να συνεχίζεται, να βρίσκει και συνέχεια. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστώ τον κύριο Λουί Γκρέκ, τον συνάδελφο, ο οποίο είχε την πρώτη ιδέα, πόσο για πρώτη φορά την ιδέα να γίνει μια μεγάλη διάσκεψη για όλα τα θέματα που αφορούν τον πολίτη τη Ευρώπη και πιστεύω ότι αυτό ουσιαστικά ήταν αυτό που πράξαμε, δηλαδή ότι εισακούστηκαν τα μελήματα, οι ανησυχίε των πολιτών της Ευρώπης, έτσι ώστε να τους δείξουμε και από πλευρά μας ότι η εσωτερική αγορά δεν είναι κάτι το ε, αόριστο, αλλά ότι τους προσφέρει προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, όπως παράδειγμα, η αναγνώριση των σπουδών, επαγγελματικών σπουδών, η δυνατότητα για σπουδές σε άλλη χώρα, πράγμα που ακόμα δεν έχει επιληθεί, ε, η ασφάλεια, η νομική ασφάλεια ως προς τις ηλεκτρονικές αγορές, δηλαδή διαδικτυακές αγορές, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλά πολλά άλλα θέματα. Πολλά ήταν τα θέματα λοιπόν που ζήτησε το φόρουμ και επισήμανε τα προβλήματα που γνωρίζουν διάφοροι τομεί τη εσωτερική αγορά. Και τώρα, κύριε Επίτροπε, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στι λύσεις που θα προταθούν. Περιμένουμε από εσά, όπως υποσχεθήκατε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνετε αυτές τις λύσεις και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και προσωπικά εγώ και η σοσιαλιστική μου ομάδα θα παρακολουθήσουμε και θα υποστηρίξουμε με εύνοια κάθε καλή πρόταση που θα καταθέσετε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκέπχαρτ και τώρα για τρία λεπτά το λόγο και ο κύριος Μπουσόη. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε Πενταλή, όπως τονίσατε επανειλημμένως, η ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς δεν πρέπει να είναι μόνο θέμα ευρωπαϊκών θεσμικών οργανών. Αυτό θα πρέπει να προκύψει από ευρύ διάλογο με τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τις εθνικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τους δικαστές και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και ήταν ε, σημαντικό και επιτυχές ε, το ε, φόρουμ ενιαίας αγοράς στην Κρακόβια και πρέπει να πω πως η συμμετοχή σε αυτό το φόρουμ ήταν πολύτιμη εμπειρία για μένα. Οι συμμετέχοντες έκαναν επικοδομητικό διάλογο που μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για το τι θεωρούν ότι είναι οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Κάτι που πρέκυψε από το φόρουμ και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι το εξής η πλειοψηφία των πολιτών και κάποιες φορές και ακόμα και μερικοί από εμά θεωρούμε ότι η νομοθεσία της ενιαίας αγοράς είναι εξαιρετικά τεχνικής φύσης και ορισμένε φορές αυτό αληθεύει. Αλλά με χαρά είδα ότι το φόρουμ προσέλκυσε πολίτες που ήρθαν για να πούν τη δική τους ιστορία σε σχέση με την ενιαία αγορά. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πως η ενιαία αγορά Καταρχήν αφορά τους πολίτες, ε, τους συλλογικούς απλούς ανθρώπους που δυστυχώς ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να χαίρουν των δικαιωμάτων τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία για την πλήρη της δέσμευση στην ενιαία αγορά και γιατί έφεραν τη δήλωση της ε, Κρακοβίας ε, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Τώρα, αν αυτό το φόρουμ, εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αποδείξουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη δήλωση της Κρακοβίας, ότι έχουμε την πολιτική βούληση να προβούμε σε αποτελεσματικές λύσεις και να τις θα πρέπει να κατανοήσουμε πως η νομοθεσία μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς όμως τη σωστή, ε, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τη σωστή και έγκαιρη της εφαρμογή σε επίπεδο 100 μελών. Θεωρώ λοιπόν πως το φόρμα αυτό είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον και είναι τρόπος για να προχωρήσουμε και σταδιακά να εξαλείψουμε τους ε, αναπομείνοντες φραγμούς και να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στην ενιαία αγορά. Γι' αυτό και στηρίζω την ιδέα του να δημιουργηθεί ένα φόρουμ online για την ενιαία αγορά, μια μόνιμη πλατφόρμα για διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους και γι' αυτό πιστεύω πως του χρόνου θα πρέπει να σηματοδοτηθεί η 20η επέτειος της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς με τη διοργάνωση παρομοίων γεγονότων εκδηλώσεων σε όλα τα κατημέλια όπως ήδη προτάθηκε. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ε, εργάστηκαν σκληρά για τη διοργάνωση του Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά, να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα τον Επίτροπο Βονταλή και Μπαρνιέ, το Κοινοβούλιο, την Πολωνική Προεδρία και όλους τους πολίτες, ε, τις επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ και όσους τους εμπειρογνώμονες συνέβαλαν στην επιτυχία του πρώτου φόρουμ για την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά τώρα, κύριο Χάρμπορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω Πρόεδρο τη Επιτροπή, θα ήθελα καταρχά ιδιαίτερω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντάλη, ο οποίο συμμετέσχε με πολύ δραστήριο τρόπο ε, στο φόρουμ και τον Επιτρόπο Μπαρνιέ βεβαίω, ο οποίο ξεκίνησε από τη Μάλτα αυτή την προσπάθεια να προσελκύσει στο διάλογο για την ενιαία αγορά ε, κάθε κράτου μέλου και βέβαια και ο κύριο Γκρέκ φαντάζομαι τον συνοδεύει. Και επίση θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ επιτυχίε ορατέ τη ε, ενιαία αγορά, του φόρουμ ενιαία αγορά και πιστεύω ότι όντω ήταν μεγάλη επιτυχία. Ε, πάνω απ' όλα διότι αποδεικνύεται ότι είναι ε, η προσπάθεια αυτή αποτέλεσμα κοινή προσπάθειας συνεργασίας εταιρική σχέσης, όχι δηλαδή ρυθμίσεις μόνο και κανόνες που επιβάλλονται από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφασίσει ένας επίτροπος μόνος του. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να, ε, να υλοποιήσει ένα κράτο μέλο δουλεύοντα μεμονωμένα. Πρέπει, όπω αναδεικνύεται να συνεργάζονται πιο καλά τα κράτη-μέλη μεταξύ τους και να στηρίζουν προς τους καταναλωτές ώστε να έχουν τις καλές υπηρεσίες, τις διαδικτυακές που και εσείς υποστηρίξατε κύριε Επίτροπε. Και πιστεύω ότι από τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε για την προαγωγή αυτού του φόρουμ ε, θα πρέπει να, να πούμε ότι δυστυχώς δεν είναι εδώ η Πολωνική Προεδρία γιατί κατέστησε ε, κύρια προτεραιότητά της αυτό το φόρουμ και εργάστηκε σκληρά για το φόρουμ για την ενιαία αγορά και μάλιστα έδωσε τις σχετικές ε, διαπιστώσεις στην ολοκλήρωση στην Σύνοδο τον Οκτώβριο, στις 23 Οκτωβρίου και πιστεύω ότι οι προσπάθειες αυτές ε, συνέβαλαν ε, τα μάλα στην επιτυχία του φόρουμ. Αλλά για να κλείνω, Πρόεδρε, το κύριο ζήτημα που παραμένει για μένα εκρεμές με, τι, με τις συζητήσεις οποίες παρακολούθησα και όπου είδαμε πόση, με πόσο ενθουσιασμό και συμμετοχή ήρθαν οι άνθρωποι, κοινοί πολίτες ε, στο φόρουμ αυτό, είναι ότι δυστυχώς λείπουν κάποιες ευκαιρίες. Δεν ήθελα επί τη ευκαιρία για να μου δώσετε και λίγο χρόνο παραπάνω Σας σα ε, συγχαρώ για την πολύ μεγάλη δουλειά που κάνατε για το διαδίκτυο που μας επιτρέπει να ενημερώσουμε τον πολίτη για την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ τον κύριο Χάρμπορ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης παρακαλώ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η μορφή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει μια αποτελεσματική ενιαία αγορά και να προσαρμόζει τις οικονομικές με τις κοινωνικές ανάγκες της αγοράς, καθώς και να ενισχύει την αλληλεγγύη, να καθιστά δυνατή την υλοποίηση των ατομικών και συλλογικών επιτευγμάτων, να συμβάλλει στην αηφόρο ανάπτυξη η πράξη για την ενιαία αγορά δεν φαίνεται όμως κατά την άποψή μας να απαντά στις σημερινές ανάγκες των πολιτών. θέλουμε να ανακτήσουμε το πλήρες και ολοκληρωμένο δικαίωμα της κοινωνίας να περνάει το δημόσιο συμφέρον πάνω από το συμφέρον των αγορών. θέλουμε να ανακτηθεί το κοινωνικό δικαίωμα να προτεύει η προστασία του πολίτη η διατήρηση των θέσεων εργασίας και οι συνθήκες εργασίας επί των κανόνων του ανταγωνισμού πρέπει να προλάβουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της κοινωνικής ευρώπης. η εναλλακτική μας πρόταση είναι απλή εύκολη και σαφώς διατυπωμένη να επικρατήσουν οι κοινωνικές ανάγκες επί των κερδών. θέλουμε να συμμεριστεί αυτή την οικονομική κοινωνική πολιτική και πολιτιστική εναλλακτική λύση ολόκληρη η ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ συνάδελφε και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, καταρχάς η κυρία Τούν Ενάμιση λεπτό Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Επίτροπο για τα πολύ φιλικά του λόγια προς εκείνους που δραστηριοποιήθηκαν, που στρατεύτηκαν για την επιτυχία του φόρουμ. Αυτό πράγματι μας έδωσε φτερά, έδωσε φτερά σε όλους αυτούς που σκληρά αγωνίζονται κάθε μέρα για να ε, καταργήσουν τους φραγμούς στην εσωτερική αγορά, στο ελεύθερο εμπόριο, στην ενιαία αγορά. Είναι κάτι το οποίο αποβαίνει όφελος και των επιχειρηματιών και των καταναλωτών πάνω απ' όλα, διότι αυτό είναι το κύριο, ε, η κύρια ομάδα, ο κύριος μοχλός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταναλωτές. Ευχαριστώ λοιπόν τον Επίτροπο Μπαρνιέ και τη Γενική Διεύθυνση Νέα Αγορά με την κυρία Γενική Διευθύντρια, τη οποία το όνομα δυστυχώ σπάνια ακούγεται, αλλά η οποία έχει συμβάλει τα μάλα στην επιτυχία αυτού φόρουμ. Ήταν μεγάλη η επιτυχία, όπω είπα, καταπληκτική εμπειρία. Και συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες ότι θα πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί ο διάλογος με την κοινωνία, με τους πολίτες, να συνεχίσουμε να εισακούμε τις φωνές ε, και τα μηνύματα που εκπέμπει η κοινωνία και πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτά τα αποτελέσματα του φόρουμ. Πόθεν, Πρόεδρε, αντλείται η επιλογή ότι το επόμενο φόρουμ θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει ληφθεί τέτοιου είδους απόφαση και αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση θα πρέπει από κοινού να τη η Επιτροπή με το Κοινοβούλιο και όχι μόνο μερός. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, ε, άλλοι χώροι που θα μπορούσε να διεξαχθεί στο επόμενο φόρμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τούν Χόνσταν, λέει ο πρόεδρος, ε, ο κύριος Κορέα Δεκάμπος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πέτρο Πεντάλη, το πρώτο φόρουμ για την νέα αγορά, η ιδέα που προκύπτει από την ε, έκθεση Γκρέχ, ε, έγινε στην Κρακοβία. Ε, πολύ καρποφόρος ήταν ε, ο διάλογος εκεί και πολύ σπουδαία η συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αλλά και της ε, κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε τις ε, στρατηγικές για τις 38 προτεραιότητες που εντοπίζονται στην ε, πράξη για την ενιαία αγορά. Αλλά για να υπάρχει αγορά χρειάζεται εμπιστοσύνη. Τώρα η εμπιστοσύνη των πολιτών και των καταναλωτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δεδομένο. Το πρέπει να τροφοδοτείται. Ε, η ενιαία αγορά είναι ένα εγχείρημα Ε, Χρειάζονται οριζόντιες πολιτικές, η υγεία, η κοινωνική προστασία των καταναλωτών, το δικαίωμα στην εργασία και η βιώσιμη ανάπτυξη. Το Φόρουμ για την ενιαία αγορά θα πρέπει έπειτα να μετατραπεί σε μια, ένα, μια εμβληματική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αιτήσια επανάληψή του και με ένα και πιο μεγάλη συμμετοχή και διάφορα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε τον κατάλογο των ομιλητών, ο κύριος Κοσούστινικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου, η ενιαία αγορά αποτελεί το μοναδικό μέσο που προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη και μπορεί να την προωθήσει περαιτέρω. Η ενιαία αγορά έχει την δική της ιστορία επί 20 και πλέον έτη και το φόρουμ στην Κρακοβία έχει επίσης ε, τη δική του ιστορία. Η αρχική ιδέα γεννήθηκε στην έκθεση Greg και εγώ ενημερώθηκα για πρώτη φορά μετά από συζήτηση με την κυρία Τούν Χώσταν και τον Μάριο Μόντι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλους τους συναδέλφους από την Επιτροπή γιατί θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία του φόρουμ αυτού και αποτέλεσε μια επιβεβαίωση για την επιτυχία αυτή το γεγονός ότι η Ρόζα Τούν χτες βραβεύτηκε ως η καλύτερη ευρωβουλευτής για θέματα ενιαίας αγοράς. Θα ήθελα να τη συγχαρώ εξ ονόματο και των άλλων συναδέλφων. Ευχαριστώ συνάδελφε Κοτσούσνικ και τώρα η διαδικασία Κάτσου. the Θα δώσω το λόγο καταρχάς στην συνάδελφο Μπατσέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ρόλο τη ενιαία αγορά είναι καθοριστικό αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει από το οικονομικό τέλμα που χαρακτηρίζει την τρέχουσα κρίση. Επίσης, χρειαζόμαστε σωστή εφαρμογή, σωστή εποπτεία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προτύπων της ενιαίας αγοράς. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς. Επίσης, τα κρατημέλη θα πρέπει να καταβάλουν πιο πολλές προσπάθειες για να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα για την ενιαία αγορά τα πλέον πρόσφατα, η χώρα μου συγκαταλέγεται στις 10 χώρες που σημείωσαν βελτίωση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με μέση καθυστέρηση 2,2 ε, μήνες ε, ε, σε ό,τι αφορά την προθεσμία εφαρμογής νομοθεσίας. Η Ρουμανία βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση είναι σαφές ότι προάγονται οι συνεργασίες μεταξύ του τοπικού, εθνικού και περιφερειακού επίπεδου για να βελτιωθεί η εφαρμογή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ενοποίηση της ε, εσωτερικής αγοράς χρειάζεται κινητικότητα, ηλεκτρονικό εμπόριο, αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο. Υποστηρίζω την πρόταση του φόρουμ να υπάρχει ένα επαγγελματικό ευρωπαϊκό φόρουμ για να προωθηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων και για να απλοποιηθεί η διαδικασία για την αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση και την απόσπαση εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη από πλευρά των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να χρησιμοποιείται το διαδικτύο. Αναμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή αγορά προκειμένου να υπάρχει αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Επίσης, χρειάζεται νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ, κυρία Τικάου. Και τώρα η συνάδελφος Γκάλμπελτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι προηγούμενοι ομιλητέ ε, μίλησαν για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τη συνεργασία. Η αναπτυξιακή, η στόχοι για την ανάπτυξη και η στόχοι για την ε, απασχόληση μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία η οποία θα πρέπει σύντομα να εξευρεθεί. Το οικονομικό όφελος ε, είναι μεγάλο και δεν θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Αλλά καταρχάς όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πληρούν και να εφαρμόσουν όλες τις πτυχές της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θα πρέπει στο σημείο αυτό να ξεχνάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ως τώρα δεν αποτέλεσαν επίκεντρο των προσπαθειών. Θα πρέπει να μειώσουμε το φόρτο που τις επιβαρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αναλάβει ως καθήκον. Αυτό και θα διεξάγει σχετική μελέτη για τα διοικητικά έξοδα. Ευχαριστώ πολύ, ο Ευχαριστώ πολύ μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίοδο κρίσης έχουμε την ανάγκη στήριξης της εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς που αποτελεί και το μεγαλύτερο παράγοντα επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποβλήθηκαν μέτρα για τη βελτίωση αυτής της ε, ενιαίας αγοράς με την ε, πράξη για την εσωτερική αγορά την οποία την οποία πρότεινε τον κανονισμό για την ιστορική αγορά που πρότεινε ο Επίτροπος Μπαρνιέ, μια σειρά μέτρων δηλαδή, στα οποία θα συνεργαστούν και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πέραν των οργάνων. Πρόκειται για μια αρχή μια αγορά στηριζόμενη στις τέσσερις ελευθερίες που λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια που όμως δεν έχει ακόμη ανοίξει πλήρως τα φτερά της, δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της και άρα τα μέτρα του κύριου Βαρνιέ είναι απαραίτητα για να επιτρέψουν σε αυτόν τον ε, τόσο σημαντικό κινητήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει πλήρη αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για να ολοκληρωθεί τώρα η διαδικασία Κατστιάη Θα λάβει το λόγο ο, Επίτροπος, ο κύριος Οτμαρκάλας. Καράς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ την κυρία Τούν για την ε, πρώτη αυτή ε, εκδήλωση του Φόρουμ για την Εσωτερική Αγορά και πρέπει να δοθεί συνέχεια. Δεν είναι έτοιμη η εσωτερική αγορά, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει κλείσει. Η εσωτερική αγορά είναι η μεγάλη δυνατότητα για την ανάπτυξη, για την εφημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προχωρήσουμε καταργώντας διατάξεις, καταργώντας απαγορεύσεις δηλαδή και φραγμούς και να και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν πλήρως, θα υλοποιούν πλήρως ε, τις διατάξεις οποίες θα εγκρίνουμε. Η εσωτερική αγορά και ένα τέτοιο φόρουμ μπορεί να αποτελέσει τον καθρέπτη στον οποίο θα αντικατοπτρίζονται κάθε έτος τα μεγάλα επιτεύγματα που οφείλουμε στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Έτσι ολοκληρώνει τη δικασία Καρστιάη. Και τώρα λαμβάνει το λόγο ο κύριος Επίτροπος, ο κύριος Δαλή. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Η συζήτηση που μόλις ολοκληρώθηκε είναι πολύ σημαντική για την ε, υλοποίηση της δέσμευσής μας να ε, προωθήσουμε την ενιαία αγορά και να ανταποκριθούμε δραστήρια στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Η επίλυση της κρίσης ε, εξαρτάται από μια αποτελεσματική ενιαία αγορά που με τη σειρά της εξαρτάται από τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τους, τους ισχυρούς καταναλωτές. Όπως είπα και στα εισαγωγικά μας σχόλια, ε, τονίζουμε την κοινωνική πτυχή της ενιαίας αγοράς, διότι δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον καταναλωτή, τον εργαζόμενο που συμμετέχουν στην αγορά. Το και στην αναρτήριά μου ε, ομιλία ότι ο στόχος είναι η προώθηση, η προόδος των πολιτών της Ευρώπης ε, και η προόδος δεν επιτυγχάνεται μέσω ενός στατιστικού μητρώου, αλλά μέσω μιας πραγματικής ποιότητας ζωής που μπορούμε να προσφέρουμε. Η αποφασιστικότητά σας για να παρέχετε στήριξη στην ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντική και όπως είπε ο κύριος Χάρμπορ και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, είναι μια προσπάθεια συνεργασίας. Πρέπει να κινηθούμε από κοινού, κράτη-μέλη, κοινοβούλιο, επιτροπή καταναλωτές, επιχειρήσεις, όλοι πρέπει να κινηθούμε από κοινού ώστε η ενιαία αγορά να καταστεί πραγματικότητα. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι 15 επίτροποι έχουμε δεσμευθεί ε, για να καλύψουμε με τις ενιαίες αγοράς ε, πολλές, ε, πολλούς τομείς και είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για την μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πάνω στο πνεύμα του φόρουμ που έγινε στην Κρακοβία. Δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο φόρουμ που διοργανώθηκε. Πιστεύουμε πως η επιτυχία του μας υποδεικνύει τη σημασία που έχει το να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα σε μόνιμη βάση και να προσπαθήσουμε να την μετατρέψουμε σε μια σειρά παρόμοιων εκδηλώσεων. Αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς τη συχνότητα με την οποία θα παραλαμβάνεται αυτή η εκδήλωση και δεν έχουμε ακόμα, κυρία Τούν, καθορίσει την τοποθεσία του επόμενου φόρουμ. Έγιναν κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν έχει λεφθεί καμιά απόφαση. Όλα είναι ακόμα υποσυζήτηση. Όπως είπαμε, από... Ούτως ή άλλως πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια και γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξει διάλογος ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε πάνω στα όσα έχουμε ήδη καταφέρει. Πρόκειται για βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για να επιτύχουμε το στόχο μας μια πολύ ενεργή και δραστήρια ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Κατ' εξαίρεση, μια και ακούστηκε το όνομά δύο φορές, ας λάβει το λόγο για άλλη μια φορά η κυρία Τσούν Ουνχόνσταν. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Ο Επίτροπος Τόντι έδωσε απάντηση στις παρατηρήσεις μου και θα ήθελα να ολοκληρώσω την προηγούμενη παρέμβαση που διακόπη για να υπογραμμίσω και αυτό που είπατε εσείς ως προς την επιλογή τη πόλη που θα δεχθεί το προσεχέ φόρουμ. Νομίζω ότι έχουμε πολλέ εκδηλώσει εδώ στι Βρυξέλλε. Αυτό το φόρουμ τη Κρακοβία στέφθηκε με επιτυχία ακριβώ επειδή ήταν έξω από τι Βρυξέλλε και έτσι μπόρεσε να διοργανωθεί κατά τρόπον ώστε να συναντήσουμε και ανθρώπους που δεν έχουμε την δυνατότητα κάθε μέρα να συναντούμε. Δέκα 10.000 πολίτες που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και που εκπροσωπούν εκατομμύρια ε, άλλων πολιτών. Σας ευχαριστώ θερμά, λέει ο Πρόεδρος. Κατατίθεται ψήφισμα πέντε ομάδων για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στι 12. Τελευταίο σημείο στην ημέρηση διάταξη για σήμερα. Έχουμε τι παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού δυνάμει του άρθρου 150 του κανονισμού με τον κύριο Τοκέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πριν από 91 χρόνια